Colleagues, Αδέλφοι, αργίζουμε την συνεδρίαση της Επιτροπής Γυναικών. Πρώτα-πρώτα, έγκριση της μέσης διατάξεως, αν δεν υπάρχει κάποια ένσταση. Δεν έχω ανακοινώσεις της Προέδρου και πάμε στο σημείο 5. Έγκριση των πρακτικών της 24ης Ιανουαρίου. Αν δεν υπάρχουν στάσεις και τα πρακτικά εγκρίνονται. Πάμε στο σημείο παριθμών 6 της ημερησίας διατάξεως που είναι τα πιλωτικά προγράμματα και προπαρασκευαστικές δράσεις του προϋπολογισμού του 2019. Η συγγήτρια για αυτά τα πιλωτικά προγράμματα είναι η Μαλίν Μπιόρκ. Αρχίζουμε την ανταλλαγή απόψεων και την αντικαθιστά την εισηγήτρια Μπιόρκ, ο κύριος Λόπες. Θα είμαι πολύ σύντομος. Η συνάδελφος δεν μπορεί να είναι παρούσα σήμερα για λόγους έκτακτης ανάγκης. Για να μας παρουσιάσει αυτά τα πιλωτικά σχέδια ζητά συγγνώμη. Έχουμε λάβει 16 προτάσεις. Θα σταλούν στην Επιτροπή ε, Προϋπολογισμού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η, η Μαλίν τουλάχιστον ευχαριστεί πολύ. Δεν έχει να κάνει σχόλια επί ε, των σχεδίων που προτάθηκαν. Μπορούμε λοιπόν να ψηφίσουμε εκτός και αν υπάρχει κάποιο σχόλιο από την δική σας πλευρά, το οποίο θα μεταφέρω στην εισηγήτρια. Thank you very much. And now I will open the floor for the, the discussion for the... Ας ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Ανταλλαγή απόψεων. Παρακαλώ, ποιος θέλει το λόγο. Ας προχωρήσουμε λοιπόν κατευθείαν στην ψηφοφορία, αφού κανείς δεν θέλει το λόγο. Please be ready for the vote. Do have... Ετοιμαστείτε, έχετε στα χέρια σας τις κάρτες, βάλτε τις στη σχισμή. Ah, okay. ah, it's not necessary to... Ah. So, um, Ας ξεκινήσουμε με τα πιλωτικά προγράμματα, σχέδια και τις δράσεις προετοιμασίας για τον ε, προϋπολισμό 2019. Υπάρχει μόνο ένα πιλωτικό σχέδιο. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Οκ, okay, ηλεκτρονική επαλήθευση αφού θέλετε έτσι. Ξεάρχεται η ψηφοφορία. Λίγη η ψηφοφορία ε, εγκρίνεται. Δεύτερο πιλωτικό σχέδιο, ποιος είναι υπέρ. Υπέρ λέω. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρίτο σχέδιο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. πληρωτικό, όχι. Ας περιμένουμε τον κύριο Ταραμπέλα. Κύριο Ρόκα. Είστε έτοιμοι. Ωραία. Υπάρχουν τέσσερα προσχέδια υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Πιλωτικό σχέδιο υπαριθμού 5. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Πιλωτικό σχέδιο 6. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Πιλωτικό σχέδιο 7. Υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. Θέλετε ηλεκτρονική επαλήθευση, ωραία, άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη. Εγκρίνεται. Πληρωτικό σχέδιο 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πληρωτικό σχέδιο 9 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται επαλήθευση και πάλι Σοβαρευτείτε παρακαλώ. Πολιτικό σχέδιο 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη. Εγκρίνεται. Πιλωτικό σχέδιο 10. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Πιλωτικό σχέδιο 11. Υπέρ. Κατά. εποχέ Εγκρίνεται. Πιλωτικό σχέδιο 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πιλωτικό σχέδιο 13 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Πιλωτικό σχέδιο 14 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Πιλωτικό σχέδιο 15 υπέρ. Υπέρ λέω. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Πιλωτικό σχέδιο 16 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Now more votes today, but we continue our farm meeting. Ωραία. Συνεχίζουμε με την υπόλοιπη συνεδρίαση μας. Uh, Το 8. Αποστολή και την εξωστή Δευτέρα Σύνοδο αφορά την Επιτροπή για την Κατάσταση των Γυναικών στη Νέα Υόρκη. Έχουμε έκθεση η οποία θεωρώ ότι εγκρίνεται αν δεν υπάρχει κάποια ένσταση. Το επόμενο. Ωραία. Συνάδελφε, ένα λεπτάκι αναμονή μια που περιμένουμε τον εισηγητή ή την εισηγήτρια. Ε, Συνάδελφοι, λέει η πρόεδρος, επειδή περιμένουμε τον κύριο Ντανιέλ Βιώτη για τον προπολογισμό και από ό,τι μα είπε θα έρθει στις 11.30, μπορείτε να ε, πάτε για ένα δεκάλεπτο διάλειμμα και αρχίζουμε στις 11.30. Συνάδελφοι, συνεχίζουμε την συνεδρίασή μα και είμαστε στο σημείο 9 Γενικός Προκουρισμός Ευρωπαϊκή Ένωση για την χρήση 2019. Όλα τα τμήματα και κεφάλαια. Ο εισηγητής μα, η εισηγήτρια καλύτερα είναι η Μάλιν Μπιόρκ. Σήμερα έχουμε ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Ντανιέλε Βιώτη που είναι συγητής για τον προϋπολογισμό. Οπότε και τον ε, δίνουμε το λόγο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και στα Ιταλικά σας ευχαριστώ όλους και όλες για την πρόσκλησή σας στην συνάντηση της Επιτροπής σας. Όπως γνωρίζετε, ως εισηγητής για τον γενικό προϋπολογισμό του 2019 παρακολουθώ τις εργασίες των Επιτροπών και ως συμπρόεδρος της ομάδας συμφέροντος για τους LGBT οπότε και είμαι ιδιαίτερος κοντά στο δικό σας έργο και στη δική σας επιτροπή. να συζητήσουμε κάποια συγκεκριμένα σημεία, αλλά πρώτα-πρώτα να δούμε με μεγάλη συντομία τα θέματα του γενικού προϋπολογισμού και τι γίνεται από του Κοινοβουλίου μας, ε, κυρίως μεθοδολογικά. Είναι το έργο μας περίπλοκο, γιατί όπως γνωρίζετε ο προϋπολογισμός είναι ένα στεγανό, κλειστό, στατικό σύστημα Οπότε και είναι δύσκολο κανείς να κινηθεί δεξιά και αριστερά, να, να μετακινήσει τα ποσά, να ε, δουλέψει εφάνταστα από πολιτικής πλευράς. Παρ' όλα αυτά το κοινοβούλιο συχνά έχει αγαθές προθέσεις και η πρόθεσή μου τέλο πάντων είναι να κάνω αυτό το οποίο έκαναν και οι συνάδελφοι τα προηγούμενα χρόνια. Να μπορέσω να συγκεντρώσω όσο γίνεται ευρύτερη συνένεση για την τοποθέτηση του Κοινοβουλίου. Και έτσι να αναζητήσουμε την συνένεση και των πολιτικών ομάδων, αλλά και να υπάρξει ευρία υποστήριξη από πλευράς των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Οπότε να μην ολοκληρωθεί το έργο μου εδώ με την συνεννόηση με την κάθε επιτροπή, αλλά να συνεχιστεί η συνεννόησή μας και για τη συνέχιση του έργου μου για τον προϋπολογισμό του επομένου έτους. Βέβαια, τώρα συζητούμε χωρίς προϋπολογισμό γιατί ακόμα δεν έχουμε το σχέδιο του προϋπολογισμού που παρουσιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε, προς το παρόν, να δούμε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές αυτές που τον Μάρτιο εγκρίναμε. Συγγνώμη για το βήκα. Τέλος πάντων, όπως γνωρίζετε έγινε η έγκριση αυτών των κατευθυντηρίων και στη συνέχεια θα συζητήσουμε για το σχέδιο προπολογισμού και θα δείτε ότι σε αυτές τις καθηγητές γραμμές έχω αναδείξει το θέμα της ισότητας των ευχηρωτήν την πολέμηση των δυσμενών διακρίσεων. Να μην πια μια παράγραφο σε μια έκθεση. Θέλω να επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε κάποια θέματα τα οποία με χαρά μου έχουν ενταχθεί στο θεματολόγιο σας και θα κρυφθούν τον πρώτο προπολισμό και αναφέρομαι συγκεκριμένα στο θέμα της επιχειρηματικότητας, της απασχόλησης και της ε, προσβασιμότητας σε δάνεια. πιο δίκαιη κοινωνία επομένω και πιο ευημερούσα. Να μπορέσουμε να φέρουμε την ανάπτυξη στην Ευρώπη. Να φέρουμε την κοινωνική ένταξη και βεβαίω πρέπει στα πλαίσια αυτά να καταπολεμήσουμε τις δυσμενείς διακρίσεις και τις διακρίσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών, τον ρωτισμό και την ξενοφοβία, την ομοφοβία, καθώς και την πρόκληση μίσους και για όλα αυτά αναφερόμαστε στην έκθεση. Και έχουμε τώρα κάποια συγκεκριμένα σημεία τα οποία ενδιαφέρουν τη δική σας επιτροπή, όπως φέρει ότι θα πρέπει να υπάρχουν κάποια χωριστά κονδύλια για το Δάφνη. Επίσης θα πρέπει να αυξηθούν για το ε, έτζε ε, οι ανθρώπινοι και οι χρηματικοί πόροι. Να καλύψουμε τις ε, πρόσφυγες και τις μετανάστες. Επίσης να δούμε τι γίνεται με τις εξωτερικές σχέσεις και να δούμε πώς η ισότητα των φύλων επίσης θα ληφθεί υπόψη στον τρόπο λειτουργία των θεσμικών οργάνων. Οπότε είπαμε θα να δούμε τι γίνεται με επιχειρηματικότητα, πιστώσεις και τι γίνεται στα πλαίσια του κόσμου του ορίζοντα 2020 αυτά τα μείζωνα προγράμματα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτω ώστε να δώσει καινούρια πνοή στην ε, οικονομία. Βεβαίως και θα ακούσω τις απόψεις σας και θέλω αυτός ο επόμενος προϋπολογισμός να είναι κάτι με το οποίο να ταυτίζονται όλοι οι Ευρωπαίοι και οι Ευρωπαίες όλοι όσοι επί χρόνια ήταν θύματα δεσμενών διακρίσεων και των κεκριμένων και των πιο φανερών. Η Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Διώτη. Και τώρα θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Πιμέντα Λόπες, ο οποίος αντικαθιστά την Μάλιν Μπιόρκ. τη εισηγήτριας τη νομοδότησής μας. Ευχαριστώ. Ήδη στο προηγούμενο σημείο της μέσης διάταξης ε, ε, είχα αναφέρει ότι η κυρία Βιόρκ δεν μπορεί να είναι παρούσα και ζητά συγγνώμη γι' αυτό. Της έτυχε κάτι απρόβλεπτο. Λυπάται πολύ που δεν μπορεί να συζητήσει με τον εισηγητή την νομοδότησή της. Η γνωμοδότηση έχει υποβληθεί προς μετάφραση. Θα συζητηθεί στην Επιτροπή μας στα μέσα Μαΐου. Η εισηγήτρια στην έκθεση αυτή αναφέρει πως οι ανισότητες είναι διαρκώς επιδεινωμένο πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο προϋπολογισμός θα πρέπει να το λαμβάνει υπόψη αυτό προκειμένου να προστατευτούν και να αναπτυχθούν τα κοινωνικά δικαιώματα ή τα, ε, οι υπηρεσίες που προσφέρονται και να έχει ως στόχο τη βελτίωση της ισότητας των δύο φύλων και την κατάσταση των γυναικών. Προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αυξήσει τη χρηματοδότηση της ε, ε, εξωτερικής ανεψυχιακής βοήθειας, ιδιαίτερα στα κεφάλαια των γυναικών και της υγείας και της παιδείας ε, και να καλύψει την ε, μείωση της συνεισφοράς στα διεθνή φόρα των ΗΠΑ. Λυπάτε, ε, τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν τα ε, ποσά του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Κοινωνικού Ταμείου για να προστατευθούν, προωθηθούν τα δικαιώματα των γυναικών μέσω της εκπαίδευσης της υγείας, ε, εκπαίδευσης ε, για τα δικαιώματα, τα παραγωγικά και σεξουαλικά δικαιώματα κλπ. θεωρεί ως προτεραιότητες για την Επιτροπή μας τα εξή. Χρήση του προπολισμού του φύλου, επεξεργασία ενός ειδικού δημοσιονομικού πλαισίου για την ένταξη του, της των φύλων στα όργανα της Ευρωπαϊκής χρηματοδότηση, επαρκή χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ισότητας των Διοφύλων, ε, ένα ξεχωριστό κονδύλιο για κάθε ειδικό στόχο του προγράμματος ε, δικαιωμάτων και ισότητας, των πολιτών, χρηματοδότηση προγραμμάτων που θα βοηθήσουν τις πρόσφυγες και τις μετανάστες να έχουν πρόσβαση στις βασικές ε, υπηρεσίες και περισσότερη χρηματοδότηση για την, βία, για την κατά των γυναικών και κατά των ΛΟΑΔ. Η κυρία Μπιόρκ ελπίζει ότι θα συνεργαστεί με ε, πολύ ε, αποτελεσματικά με την Επιτροπή Προπολογισμών και με τα μέλη της Επιτροπής Γυναικών. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ε, η Πρόεδρο. σας ευχαριστώ και εγώ κύριε Λόπες. Τώρα, να δώσουμε το λόγο στους κυρίους συγητές και πρώτα η κυρία Μόνικα Βάνα. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους δυο σας για τις εισαγωγικές παρατηρήσεις, ιδίως τον κύριο Βιώτη που ήρθε σήμερα στην Επιτροπή Δικαιωμάτων Γυναικών. Για τους πράσινους τα πιο σημαντικά ή το πιο σημαντικό κάθε φορά είναι το, ε, τα κονδύλια του προπολογισμού για την ισότητα των φύλων, που αποτελεί και υποχρέωση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι απογοητευτικό για όλε εδώ εμά, ιδίω τη Επιτροπή Δικαιωμάτων Γυναικών, που δεν συμβαίνουν τόσο πολλά πράγματα όσα θα θέλαμε εδώ και χρόνια. Διότι, όπω είπα, είναι και υποχρέωση τη Ένωση να εφαρμόσει το gender mainstream και στον προπολογισμό. Από τα πιο σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τη δική μας εδώ Επιτροπή Δικαιωμάτων Γυναικών σε ό,τι αφορά τα όσα είπατε υποστηρίζουμε όλα όσα είπατε και οι δυο σας. Ίσως να πρέπει, έχοντας υπόψη και το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, να πρέπει να τονίσουμε ότι χρειαζόμαστε μια βαθιά αλλαγή του προπολογισμού να περάσει σε ένα σύστημα ιδίων πόρων. Αυτό θα προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα. Και όπως είπατε, τα μεγάλα σημαντικά ταμεία, η ΕΣΕΦ, ΕΦΡΕ κλπ. να που θα μπουν και στη συζήτηση για την περιφερειακή πολιτική να περιλάβουν και κάποια άσκηση κριτική. και για το F-Site, για, για, για, για το EFSI, για το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, που εκεί δεν γίνεται καμιά σχετική επένδυση για τα θέματα που λέμε. Αυτά θα ήθελαν να περιλάβουν οι πράσινοι και μέσω τροπολογιών δηλαδή μεταξύ και των υπολείπων που έχετε ήδη αναφέρει. Ανεξάρτητο κονδύλιο, για παράδειγμα, για το πρόγραμμα DAFNE και αύξηση των σχετικών προβλέψεων, κάτι που ζητούμε κάθε χρόνο. Και ο δεύτερος ε, από εσά είπε να καλυφθεί το κενό που αφήνουν οι, ε, οι Ηνωμένε με την απόσυρση της χρηματοδότησής τους. είναι κάτι το οποίο απασχολεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και το βρίσκει ως στόχο και που το είδαμε και στην αποστολή στη Νέα Υόρκη ότι εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει σημαντικό ρόλο για το κλείσιμο του κενού μετά από τις δραματικές αυτές αλλαγές της αμερικανικής πολιτικής. Είναι λοιπόν πράγματα τα οποία μπορούμε να τονίσουμε ιδιαίτερα στην γνωμοδότηση. Ε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος. Η ε, κυρία Πιτσέρνο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ να ευχαριστήσω και να πω μπράβο στον κύριο Βιώτη για τη δουλειά του. Για την ευαισθησία που έδειξε για το πόσο πρόσεξε τα θέματα της Επιτροπής μας. Αυτό απορρέει αβίαστα από τις κατευθυντηρίες γραμμές. Είναι πολύ σημαντική η συνεργασία μας μαζί σας και βέβαια θα είναι και καρποφόρα και θα αποδώσει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Λαμβάνοντα επίση υπόψη, αυτό το πήρε ο κύριο Λόπε, ο μίλησε στη θέση της ε, κυρίας κυρία ε, Μπιόρκ. Θέλω να πω για το Δάφνη. Όπω γνωρίζετε και το είπαν και οι προλαλήσαντε, υπήρχε και σε παλιούς ε, προϋπολογισμούς είναι σημαντικός ως στόχος το πρόγραμμα αυτό αφορά την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά της γυναίκας ε, σε δημόσιο χώρο και στο σπίτι και επίσης στο δουλεμπόριο και από το 2014 αυτό το πρόγραμμα ε, έχει ενταχθεί στις αντίστοιχες πολιτικές και όπως ήδη είπατε θα πρέπει να έχουμε για το Δάφνη ένα χωριστό κονδύλιο και όχι μόνο για να αυξηθεί η πρικοδότηση αλλά για να αναδειχθεί η προτεραιότητα και η σημασία του προγράμματος αυτού. Και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται, τι πόρτια από την Ευρώπη για την ισότητα των ε, φίλων. Όπως είπαμε είναι θέμα αναπαραγωγικών δικαιωμάτων, θέμα υγείας, και άρα χρειάζεται χρηματοδότηση για να μπορέσουμε να ε, διαχειριστούμε αυτά τα θέματα και να καταβληθεί και πάσα δυσμενής διάκριση. Και ε, βέβαια έχω να πω ότι είναι εγκάρσιο οριζόντιο αυτό το θέμα γι' αυτό και θα πρέπει τα διορθωτικά ταμεία, η έρευνα, ε, να αποτελέσουν κομμάτι της μεθοδολογίας μας. Η χειραφέτηση της γυναίκας, όπως και εσείς είπατε στην αρχή κύριε Βιώτη, θα πρέπει να συνεχίσει να οδηγήσει στην οικονομική χειραφέτηση που είναι κάτι το βασικό και άρα να, κάτι να γίνει για την απασχόληση, γιατί η δουλειά σημαίνει ανεξαρτησία για τη γυναίκα. Και επίσης θεωρώ ότι το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης θα πρέπει να συνεχίσει την υποστήριξη σε πάσα επένδυση για τη φροντίδα των προσώπων, για τους ανηλίκους, για τους υπερηλίκους κλπ. Όλα, όλα αυτά τα οποία είναι στάδια της ζωής της γυναίκας. Επίσης για, για το μεταναστευτικό, για την ασφάλεια, για την ανάπτυξη όπου η ισότητα των φίλων είναι για όλα αυτά σημαντική. Επίσης, το είπαμε και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές στο Κοινοβούλιο, το θέμα της συγκεκριμένης υποστήριξης για τις γυναίκες που αιτούν άσυλο. Γιατί εκεί υπάρχει διαφορετική διάσταση, υπάρχουν ιδιοτυπίες, ιδιομορφίες σε σχέση με τους ε, άντρες. Έχουμε ζητήματα εκμετάλλευσης και εν μπορούμε να πούμε ότι είναι πάρα πολλά τα ζητήματα τα οποία αξίζουν τις ιδιαίτερης προσοχής μας. Οπότε θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στα θέματα της γυναίκας. Οπότε έτσι αυτό σημαίνει ότι κάνουμε βήματα πρόοδου. Και όπως είπα στην αρχή προσδοκούμε μια συγκεκριμένη συνεργασία και το ελπίζουμε θα γίνει έτσι γιατί ξέρουμε την ευαισθησία σας. Thank you. Thank you very much. Ευχαριστώ. Ο λόγος στην κυρία Ζαμπόρσκα. Καταρχήν δεν είχα σκοπό να πάρω το λόγο, αλλά θέλω να ευχαριστήσω την, τον εισηγητή Το κύριο Βιώτη που μας παρουσίασε τη φιλοσοφία του σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό. Έγινε λόγος για το πρόγραμμα Δάφνη. Η ερώτησή μου είναι πώς είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη να χρηματοδοτεί τον τρίτο κύκλο του προγράμματος Δάφνη με παραπάνω από 500 εκατομμύρια χρηματοδότηση ως τώρα και πριν από μία ώρα εδώ ακριβώ συζητούσαμε την σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και αναφέραμε ότι η βία κατ' γυναικών και η οικιακή βία αυξάνονται. Εμείς χρηματοδοτούμε τόσα χρόνια το πρόγραμμα Δάφνη και η οικιακή βία αυξάνεται. Θα ήταν πιο εύκολο να εγκρίνουμε μια περαιτέρω χρηματοδότηση αν είχαμε μια αξιολόγηση των τριών κύκλων του προγράμματος Δάφνη. Να βλέπαμε τι αποτελέσματα έχει δώσει το πρόγραμμα αυτό και γιατί χρειαζόμαστε επιπλέον χρηματοδότηση. Το να ζητάμε περισσότερα χρήματα χωρίς μελέτη ε, είναι αβάσιμο. Ίσως δεν ζητάει τη δική μου γνώμη ο εισηγητής, αλλά να πρότεινα να ζητούσαμε από την Κομισιόν να αξιολογήσει τα πάνω από 15 χρόνια λειτουργίας του προγράμματος Δάφνη. Ευχαριστώ. Κυρία Νόιχελ. Ούτε και εγώ είχα σκοπό να ε, λάβω το λόγο, αλλά η δική σας κυρία Ζάμπορσκα οδηγεί στην δική μου. Είναι σφάλμα να αμφισβητηθεί η αξία του προγράμματος Δάφνη. Χρειάζεται ένας κοινοτικό προπολογισμό που να έχει καθαρά το στόχο να προωθήσει την ισότητα και μέσω των κονδυλίων γιατί αλλιώ προγράμματα μόνο για την αντιμετώπιση της βίας είναι μόνο τα, είναι μόνο τα ψίχουλα, ενώ τη μερίδα του λεόντος λαμβάνουν τα υπόλοιπα προγράμματα. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το σημαντικό και ε, πρόγραμμα το οποίο έχει αποδείξει την αξία του, η Δάφνη δηλαδή, χρειάζεται να ενισχυθεί. Αν ξεκινήσουμε καινούργια προγράμματα, χρειάζεται πρώτα αυτά να γίνουν γνωστά και μετά να αρχίσουν να απορροφώνται τα κονδύλια τους. Εμείς οι γυναίκες θέλουμε και εμείς επιτέλους ένα τμήμα από τη μερίδα του λέοντος. Και γι' αυτό χρειάζονται περισσότερα χρήματα στον τομέα αυτό. Και ούτως ή άλλως βέβαια σε όλα τα κονδύλια, διότι μιλούμε εν τέλει για το 52% του συνολικού ευρωπαϊκού πληθυσμού που είναι γυναίκες και να αναρωτηθούμε οι πόροι που καταλήγουν, καταλήγουν σε άδικη κατανομή. Γι' αυτό και έχουν δίκιο οι προλαλήσαντες ότι πρέπει να συνεχίσουμε και να ρίξουμε γενναιόδωρα κονδύλια στο πρόγραμμα Δάφνη. Ευχαριστώ λοιπόν. Αυτά ήθελα να Άννα Ζαμπόρσκα θέλετε να πείτε κάτι ακόμα. Ευχαριστώ, λέει η κυρία Ζαμπόρσκα. Ευχαριστώ τη συνάδελφο κυρία Νόιχελ. Αν όμω είχε προσέξει καλά τι είπα, θα άκουσε ότι εννοώ το ίδιο όπως και η ίδια. Εγώ όμως θα ήθελα εκτός αυτού να έχουμε στα χέρια μας μια μελέτη που να μου δείξει ότι οι πόροι του προγράμματος Δάφνη έχουν διατεθεί σωστά και ότι δεν περικόπτονται. Αυτό εννοούσα. Να μπορούμε να αποδείξουμε ότι χρειαζόμαστε και περισσότερα ακόμη κονδύλια. Σας ευχαριστώ. Τώρα, για τα συμπεράσματα ο κύριος Δανιέλε Βιώτη που είναι ο εισηγητή του προπολισμού, για να εξαγάγει τα συμπεράσματα. Ακτό το καλύτερο κατά κάποιο τρόπο γιατί το όνομά σας ε, είναι το θηλυκό του δικού μου. Τέλος πάντων είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Ευχαριστώ όλους όσους συνέβαλαν και για όλα αυτά τα οποία άκουσα έχω να πω μόνο ότι συμφωνώ. Και προσπάθησα δύο λίγων να σας πω τι έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό σε σχέση με τις κατευθυντήριες γραμμές, τις ε, προοπτικές που εγκρίναμε τον Μάρτιο. Άκουσα και τον συνάδελφο Πιμέντα, εξ ονόματος της συγγήτριας, άκουσα και την κυρία Βάνα και θέλω τους συναδέλφους και τις συναδέλφες να τους καθησυχάσω. Ε, τα είπαμε και στην Επιτροπή των Προϋπολογισμών. Και εκεί πέρα ε, τα λέμε επίσης και τους έχω καλύψει ε, σε σχέση με τις επιφυλάξεις του. Πάντως όσον αυτό το επόμενο δημοσιονομικό πολιετές πλαίσιο θα συνεργαστούμε τους αμέσχουμους μήνες και εγώ θεωρώ ότι θα πάμε για μείζωνα μεταρρύθμιση και θα είναι ε, θαραλέα η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όχι μόνο ποσοτικά και ποιοτικά. Οπότε θα υπάρξει ευξημένη ποιότητα σε αυτό το πολιτες πλαίσιο που θα το προσδώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα είναι και το θέμα των νέων ιδίων πόρων. Και σήμερα το πρωί ε, είπαμε ότι θα πρέπει να έχει τη η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανακτήσει κάποιους πόρους, να ξέβρεται πούμε, κάποιους πόρους για τις ε, πολιτικές. Τώρα Όσον αφορά τα όσα άκουσα στις παρεμβάσεις σας και συγκεκριμένα άκουσα την κυρία Πιτσέρνο, την κυρία ε, Νόχελ, την κυρία Ζαμπόρσκα και επιτρέψτε να σας πω ότι εστιαστήκατε σε κάτι που δεν είναι ποσοτικό, είναι πολιτικό το ΣΥΠΗΝ. Και τελικά όλοι, όλοι στο ίδιο το, το πήγατε, το ότι είναι, έχει σημασία ένα πρόγραμμα που θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί πέραν των επιδόσεων του προγράμματος, πέραν των αποτελεσμάτων, γιατί έχει συμβολική, είναι εμβληματικό όσον αφορά την καταπληκτική της βίας, την ισότητα των φίλων κλπ. Και συμφωνώ ότι πολύ ε, συχνά κολλάμε στο ποσοτικό θέμα. Και είναι προφανές από τη στάση του κόσμου αν αποδίδει ένα πρόγραμμα ή όχι. Οπότε όντω και πέραν των αριθμών ή των ποσών θα πρέπει να υπάρχει υποστήριξη ενός προγράμματος από πολιτικής πλευράς επίσης. Α, όπως το είπαμε και στο κείμενο, είναι και αυτό το οποίο είπατε και μια φορά ως Ιταλό ε, το πώς ο προπολογισμό θα καλύψει τις ε, γυναίκες που είναι πρόσφυγες και που ετούνται ασύλο. Την Ιταλία προέρχομαι και ξέρετε. Και εσείς κυρία Πιτσέρνο. Το πόσο κοντά είμαστε, το πόσο έχουμε άμεση εμπειρία, όπως και τόσοι άλλοι στην Ευρώπη, το πόσο ε, πόσους κινδύνους διατρέχουν αυτές οι γυναίκες που έρχονται στην Ευρώπη και υπάρχουν κινδυνοί και στο ταξίδι που κάνουν αλλά και όταν φτάνουν εδώ και κοντά στο σπίτι μου στη Βεντιμίλια εκεί έχουμε αρχίσει να ερευνούμε για κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει και ποια αφορά αυτό την παρενόχληση των ε, γυναικών στα κέντρα υποδοχής. Αυτό το φαινόμενο εξελίσσεται εδώ και κάποιους μήνες. Άρα θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ασχοληθεί και με αυτό. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή στη συζήτηση, για την έκθεσή σας και θέλω να έχουμε έναν ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας μέχρι και την έγκριση του προϋπολογισμού. Η Πρόεδρος. Ευχαριστώ αγαπητέ ε, κύριε Βιώτη για την παρουσίαση των βασικών προτεραιοτήτων του Κοινοβουλίου για τον προπολογισμό του επομένου έτους. Ελπίζω ότι δεν θα λησμονήσετε τις προτάσεις που θα σας υποβάλει η Επιτροπή Δικαιωμάτων Γυναικών και σας εύχομαι βέβαια καλή επιτυχία στην σύνταξη του προϋπολογισμού. Σας ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφοι, πάμε στο σημείο 10 της ημερησίας διάταξης. Μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ε, σεξουαλικής και ηθικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας. Στους δημόσιους χώρους και στην πολιτική ζωή της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, η συγγήτρια είναι η κυρία Πιτσέρνο. Θα της δώσω το λόγο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρόκειται για αυτή την χάραξη κάποιες στρατηγικές για την παρενόχληση στο σπίτι και σε δημόσιο χώρο των γυναικών και τα έχουμε πει πολλές φορές για το θέμα αυτό και τα στοιχεία και σε περιφερειακό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναδεικνύουν αυτό το πρόβλημα το οποίο είναι ανησυχητικό. Οπότε και θα πρέπει να χαράξουμε μια στρατηγική πρόληψης και ανάσχεσης του προβλήματος με κάποιο δόκιμο, αποδοτικό τρόπο. Και οι τρόποι αυτών των ενοχλήσεων, των παρενοχλήσεων αλλάζουν, εξελίσσονται. Να θυμάμαι τώρα το, το, το μη του το οποίο ε, περιχαράκωσε με καινούργιο τρόπο το θέμα το θέμα της παρενόχλησης και θα πρέπει να εξεύρουμε και διάφορους πόρους διαφορετικού είδους, γιατί το θέμα είναι αντίστοιχα περίπλοκο. Ακριβώς γιατί οι μορφές της παρενόχλησης αλλάζουν και εξελίσσονται. Α, και κατανό έχω τις νέες τεχνολογίες. Και τελικά τα πράγματα βέβαια είναι ιδιαίτερα απειλητικά με συγκεκριμένο τρόπο. Οπότε έχουμε τώρα και πέραν των κλασικών και καινούριου ασύνθεστου ε, τρόπου παρενόχληση και έτσι επιβάλλεται να βρούμε κάποιου τρόπου, κάποιε στρατηγικέ ε, για να ε, σταματήσουμε αυτή την εξέλιξη. Η στατιστική είναι ξεκάθαρη. Πάνω από μία στις δύο γυναίκες είναι θύμα βίας και παρενόχληση στην Ευρώπη. Και αυτό σε οποιαδήποτε στιγμή, σε οποιαδήποτε κατάσταση, σε οποιαδήποτε χώρο. Όμως δεν υπάρχει αντίστοιχος ε, τόπος, αντίστοιχο βήμα όπου να μπορεί να καταφύγει η γυναίκα. Βέβαια άσυλο είναι, ή θα έπρεπε να είναι η τύχη του σπιτιού, αλλά και εκεί πολλές φορές το σπίτι γίνεται παγίδα από την οποία είναι δύσκολο να δραπετεύσει κανείς. Επίσης και σε δημοσιοχωρή δύσκολη η θέση της γυναίκας και στο σινεμά, στο χώρο δουλειά στο μπαρ. Οπότε, πάντως σε όλο τον κόσμο, όπως ξέρουμε, αυτά συμβαίνουν. σε μερικές χώρες τώρα ξεκίνησε αυτή η κατάσταση, αλλά βλέπουμε ότι έχουμε και την ηθική παρενόχληση, το mobbing, οπότε αυτό καταλήγει σε μια κατάσταση διάκρισης αλλά που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και με αυτόν τον τρόπο, από αυτή την οπτική γωνία οπότε. Πρόκειται για μορφές βίας που χαρακτηρίζουν και τις πατριαρχικές δομές της κοινωνίας αλλά και είναι ένας νέος τρόπος αντίδρασης στην ε, χειραφέτηση των γυναικών. Καταπολέμηση που μας χρειάζεται και στιγματισμός τέτοιας βίας. Και όπως έλεγα στην αρχή, υπάρχει σήμερα και από κοινωνίας μια καινούργια αντίληψη για το τι θα πει παρενόχληση. Και είναι και νομικό το θέμα και αυτό είναι το πιο σημαντικό πρέπει να αναδείξουμε κατά τη γνώμη μου. Και ακόμα έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας γιατί είπαμε είναι και θέμα κοινωνικό και είδατε τον τελευταίο καιρό με το μη του τι θέματα αναδείχθηκαν τι πάει να πει δηλαδή παρενόχλησε οπότε τελικά όμως όλα αυτά δεν κατέληξαν σε κάποιον νομικό ορισμό της ε, παρενόχλησης. Όλα αυτά μειώνουν βέβαια τις γυναίκες και θα πρέπει να υπάρξει παραδοχή ότι υπάρχει ισότητα ανδρών και γυναικών. Τα έχουμε πει τόσες φορές στην Επιτροπή μας και το επαναλαμβάνω ότι είναι και πολιτιστικό το θέμα και γι' αυτό πρέπει να ενεργήσουμε. Να σταματήσει η αναπαραγωγή αυτών των τοξικών στερεοτύπων. Και δεν θυμάμαι σε ποια ολομέλεια Στρασβούργου ή Βρυξελών ακούστηκαν απαράδεκτα πράγματα. Τα είπανε συνάδελφοι, ε, θεωρώντας ότι η γυναίκα είναι κατώτερο συναδελφοι είναι κάποιο είδους υποκουλτούρας. καποιο εκεί βγαίνουν οι δυσμενείς διακρίσεις των οποίων εμείς κάθε μέρα είμαστε θύματα. Και επίσης από εκεί ε, προέρχονται οι παρενοχλήσεις, αλλά δεν είναι μόνο αυτό η συνέπεια. Είναι και ότι γενικότερα τίθεται να η αξιοπρέπεια της γυναίκας σε κάθε τομέα της ζωής. Είναι πολύ σημαντικό για το τι θα κάνουμε η παιδεία. Στην παιδεία θα πρέπει σε όλες τις φάσεις του να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα από τον παιδικό σταθμό μέχρι το πανεπιστήμιο και άρα με την μελέτη αυτή που συζητούμε εδώ στο Κοινοβούλιο, όταν ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος, αυτή η διαδρομή, θα πρέπει να βρούμε και εμείς έναν ορισμό για αυτά τα φαινόμενα, γιατί δεν υπάρχει ομοιογένεια στην αντιμετώπιση, στην αντίληψη σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να έχουμε κάποιο συγκριτική ανάλυση του φαινομένου. Και στις πιο σοβαρές, πιο βαριές περιπτώσεις ε, παρενόχλησης βλέπουμε ακόμα και όταν θύματα είναι ανήλικοι, ακόμα και τότε ε, δεν υπάρχει ομοφωνία για, την, για, τη σύλληψη του τι, τι είναι αυτό το φαινόμενο. Άρα χρειαζόμαστε κοινό πανευρωπαϊκό ορισμό του φαινομένου. Πολύ σημαντικό. και για το φαινόμενο σε δημόσιο χώρο, οπότε θα πρέπει να καλύψουμε κάθε χώρο και ιδιωτικό. Να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη της τεχνολογίας που έχει δημιουργήσει νέους δημόσιους χώρους. Άρα δεν υπάρχει τελικά αρκετός έλεγχος, δεν μπορεί να υπάρξει και είναι άπειροι πια οι χώροι που μπορεί να γίνει κάτι που είναι δημόσιο και μιλώ για το ίντερνετ και τα μέσα κοινωνική δικτύωσης. Και επίσης η ρηματική ε, παρενόχληση πρέπει να μπει στον ορισμό. Έχουμε πάρα πολλές ε, περιπτώσεις εκδίκησης μέσω πορνογραφικού υλικού. Και όλα αυτά γίνονται με το facebook, με το twitter, με τα διάφορα messenger και όλα αυτά έχουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα που είναι ισοπεδωτικό για τη ζωή μιας γυναίκας. Πολλές αυτοκτόνησαν γιατί θεώρησαν ότι η αμάβρωση του προσώπου τους είναι ανέκλητη. Δεν θα πρέπει να περιοριστούμε και να δούμε πώς θα συνδυαστεί η προσπάθεια μας αυτή με την αντιμετώπιση από πλευράς των δικαστηρίων. Να μην καταλήξουν με την προσπάθειά μας ακόμα πιο απομονωμένες οι γυναίκες. Έχουμε επομένω το μόμπινγκ, την παρενόχληση στην Ευρώπη. Ε, υπάρχει ποικιλία αντιμετώπισης και αντίληψης. Προς αυτήν την κατεύθυνση πήγε η Επιτροπή Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, οπότε τελικά να έχουμε κάποια μέσα πολιτικής, τα οποία να είναι υποχρεωτικού χαρακτήρα και αποδοτικά. Οπότε με τέτοιου είδους μέσα πολιτικής και νομικής φύσης μόνο έτσι θα βρούμε την δύναμη που χρειάζεται για να ανασχέσουμε αυτό το φαινόμενο στους δημόσιους χώρους. Να λάβουμε υπόψη ποια είναι η άριστη πρακτική όπου υπάρχει, ποια είναι τα πιο αποτελεσματικά μέσα και να υπάρχει τελικά νομοθετικό πλαίσιο δεσμευτικό για να υπάρξει αντιμετώπιση και η πρόληψη. Μια αποφασιστικότητα θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή τη διαδρομή της ε, ισότητας οπότε θα πρέπει να υπάρχει και προλήψη και καταστολή να μειώσουμε τις περιπτώσεις παρενόχλησης και μόμπιν ότι υφίστανται οι γυναίκες κάτι το οποίο είναι προτεραιότητα για την Επιτροπή μας αλλά θα έπρεπε να είναι και προτεραιότητα για όλη την Ένωση. Η Πρόεδρος, σας ευχαριστώ κύριε Θα δώσω το λόγο τώρα στην σκιώδη συγγήτρια κυρία Ζαμπόρσκα εξ ονόματος του Λαϊκού Κόμματος. Ευχαριστώ πολύ αγαπητή Πρόεδρε. Ευχαριστώ βεβαίως και την εισηγήτρια για την εισαγωγική της τοποθέτηση. Νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε όλες οι παρούσες εδώ ότι η γενετήσια παρενόχληση και η ηθική παρενόχληση, το mobbing είναι σαφέστατα ένα πρόβλημα. Ότι δεν μπορούμε να το αγνοούμε το πρόβλημα αυτό. Η Επιτροπή μας έχει σκοπό να συντάξει σχετική έκθεση και αυτό αποτελεί από μόνο του απόδειξη του πόσο σοβαρά λαμβάνουμε υπόψη μας το θέμα αυτό. Πρόκειται για πρόβλημα και με ευνηδιάζει το γεγονός ότι στη σημερινή, στη σύγχρονη κοινωνία και στη σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι προηγμένη και η οποία είναι και προηγμένη και οικονομικά. Παρ' όλα αυτά, η αρνητική αυτή πτυχή, η αρνητική αυτή εξέλιξη επιμένει και υπονομεύει την ε, ισότητα ανδρών και γυναικών ερχόμενη σε αντίθεση με την ίδια την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τον σεβασμό που της ανήκει. Και αυτό έρχεται σε αντίθεση με όλα με όλες τις συμβάσεις και συνθήκες που έχει υπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν ώψη των πλέον πρόσφατων εξελίξεων, τίνω να θεωρήσω ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα το οποίο θίγει ολόκληρη την κοινωνία με πώς δεν ε, μας απασχολεί περισσότερο. Αρχίζει και μας απασχολεί τώρα περισσότερο, διότι βεβαίως μιλούν περισσότερο τα θύματα. Ε, θύματα τα οποία μέχρι πρόσφατα ε, δίσταζαν, έκρυβαν το γεγονός ότι έπεφταν θύματα παρενοχλήσεων. Δεν δημοσιοποιούσαν την κατάσταση αυτή. Από την άλλη μεριά η κοινή γνώμη καθίσταται ε, πιο ευαίσθητοι και πιο συνειδητοποιημένοι απέναντι στο πρόβλημα. Το μόμπινγκ και η γενετήσια, η σεξουαλική παρενόχληση δεν είναι και κάτι το ε, normal, είναι κάτι το αρνητικό. Ε, είναι ένα είδος άσκησης βίας και θα πρέπει να αντιταχθεί κανείς, διότι είναι άσκηση βίας σε βάρος προσώπων, τα οποία είναι θύματα. Σας ευχαριστώ και για τη μελέτη που ανετέθη και συντάχθηκε και τι μπορεί να κάνει κανείς τώρα, θα με ρωτήσετε, ώστε τα ίδια αυτά παρενοχλήσεων να αντιμετωπιστούν και ε, ιδεωδώς να εξαλειφθούν από την κοινωνία. Ε, κάνει συγκεκριμένες ορισμένες παρατηρήσεις και την ευχαριστώ για, αυτή, για αυτό και ορισμένες συστάσεις. Εμείς βεβαίως ενθαρρύνουμε με τη σειρά μας τα θύματα να καταγγέλουν τις ε, πράξεις αυτές, όμως μεγάλη σημασία έχει το επόμενο βήμα μετά την καταγγελία. Από τη στιγμή δηλαδή που το θύμα ε, καταγγέλει την πράξη, χρειάζεται να λάβει υποστήριξη, ηθική υποστήριξη, αλλά και υποστήριξη αντικειμενική υπό την έννοια του δικαίου. Όσο δεν υπάρχει η νομική προστασία, η οποία μάλιστα θα πρέπει να είναι ε, δωρεάν, θα πρέπει δηλαδή να την εγγυάται το δημόσιο, ε, δεν θα προχωρήσουμε. Γνωρίζουμε ότι στις χώρες εκείνες όπου σημειώνεται διάκριση στον τόπο εργασία, όπου υπάρχουν και οι ανισότητες αμοιβών στον τόπο εργασία. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι εκεί όταν σημειώνονται παρενοχλήσεις στον τόπο εργασία. Όταν μετά την καταγγελία παρεμβαίνει το κράτος και υποστηρίζει το θύμα, μειώνονται οι περιπτώσεις αυτές παρενοχλήσεων. Όταν όμως το θύμα γνωρίζει ότι το κόστος και ενδεχομένω και την δικαστική δαπάνη θα κληθεί να την φέρει το ίδιο το θύμα, τότε θα διστάσει ακόμα περισσότερο να ε, καταγγείλει δημόσια τις πράξεις αυτές. Είναι διαφορετική κατάσταση ανά χώρα μέλο. Αν δει κανεί τι γίνεται και πόσο συχνέ είναι οι παρενοχλήσει και κάνει τη σύγκριση μεταξύ των ετών 2010 και 2015, δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ αυτή η σύγκριση, αλλά εάν εξετάσει κανεί τα στατιστικά στοιχεία, βλέπει ότι οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης αποφεύγουν από οι παλαιέ χώρε μέλη. Σε σύγκριση με τις νέες χώρες την περιπτώσει και εδώ αναφέρονται ιδιαίτερα η Βουλγαρία και η Πολωνία και, και βλέπετε και ποιες χώρες είναι στις ε, δυτικές χώρες μέλη. Εκεί ίσως η Ιταλία ε, είναι εξαίρεση. Διαπιστώνει κανείς ότι στις δυτικές χώρες ε, είναι πολύ περισσότερες οι πανοχλήσεις από τις ανατολικές. Δεν εννοώ ότι είναι σπανιότερες οι περιπτώσεις ε, που εκδηλώνονται παρενοχλήσεις ηθικού χαρακτήρα ή ε, ε σεξουαλικού είναι λιγότερες στην ε, Ανατολική Ευρώπη, αλλά ίσως γίνονται περισσότερο ανεκτές στη Δυτική. Οι ορισμένες παρενοχλήσεις δεν χαρακτηρίζονται ως τέτοιες. Αυτό εννοώ ότι στις δυτικές χώρες, με αυτόν τον τρόπο δηλαδή ε, θεωρώ ότι στις δυτικές χώρες ε, υπάρχει μεγαλύτερη ε, ας πούμε διάδοση και υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις δυτικές και ανατολικές ευρωπαϊκές χώρες. Και κάτι άλλο, ειδικά εδώ για την Επιτροπή Δικαιωμάτων Γυναικών θεωρώ ότι έχει σημασία. Δεν ξέρω αν έχει κανείς πληροφορίες σχετικά με το τι γίνεται με mobbing και sexual harassment σε βάρος ανδρών. Δεν βρήκα τίποτα σχετικό στην μελέτη. Τι γίνεται αναλογικά ε, μεταξύ ανδρών και γυναικών οστήματα θύματα πάντοτε. Είμαι βεβαία ότι είναι λιγότερε περιπτώσει παρενοχλήσεων σε βάρο ανδρών. Ωστόσο, συμβαίνουν και αυτά. Και ε, ηθική αλλά και γενετήσια παρενόχληση και σε βάρο ανδρών. Εν πάση περιπτώσει, ε, αναμένω με ενδιαφέρον την έκθεση και εξ ονόματος του κόμματός μου, του Λαϊκού Κόμματος, σας δηλώνω ότι θα συνεργαστούμε για την σύνταξη της έκθεσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Πρόεδρος. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εμπειρογνώμονα, καθηγητή Χέλγε Χουλ, για να παρουσιάσει την μελέτη που ανέθεσε το τμήμα πολιτικής για τα δικαιώματα των πολιτών και για συνταγματικά θέματα. Κύριε Καθηγητά, έχει το λόγο. Ευχαριστώ για αυτήν την ευκαιρία. Θα ήθελα εισαγωγικά να πω ότι το πεδίο αυτής της έκθεσης είναι αρκετά ευρύ. Εστιάζεται σε διάφορα ζητήματα σχετικά ε, για το χώρο εργασία, στους δημόσιους χώρους και στην πολιτική ζωή ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα τα δούμε χωριστά, αλλά σχετίζονται μεταξύ τους. Αυτά που ισχύουν για ένα από αυτούς τους χώρους ισχύουν σε μεγάλο βαθμό και για τους υπόλοιπους. Είναι βέβαια λίγο παράξενο εγώ που είμαι σχετικά ηλικιωμένο να κάνω αυτή την παρουσίαση. Ίσως θα έπρεπε να την κάνει μια νεότερη γυναίκα, αλλά εν πάση περιπτώσει έχω εργαστεί σε αυτό το, θέμα εδώ και πολύ καιρό. Okay. Yeah, I make a sign. I just okay. So. Sorry about this. We'll go on. It's just uh, handy to have them. So if we can move on to third. Ποιοι ήταν οι στόχοι της μελέτης αυτής. Είναι να καταγράψουμε όλα τα θέματα τα οποία εξετάζουμε εστιάζοντας στα βασικά πορίσματα έρευνας και νεότερων συζητήσεων. Θέλουμε να εντοπίσουμε τι έρευνε, ε, ε, τα ισχυρά σημεία και τι αδυναμίες, καθώ επίσης και τι τάσει που εντοπίζουν αυτές οι μελέτε και τι βασικέ δράσεις τι οποίες ε, θέλουμε να αναλυθούν με τις αδυναμίες και τα ισχυρά του σημεία. Ξεκινάμε λοιπόν με κάποιες διευκρινήσεις όρων. Σε διεθνείς όρους το τι θεωρείται ε, παρενόχληση, ηθική παρενόχληση, μόμπινγκ, bullying κλπ. Ε, ε, συγκλίνουν σιγά σιγά. Και τώρα πια συμφωνούμε αρκετά. Όταν μιλάμε για bullying, είναι, μιλάμε για την έκθεση για μεγάλο διάστημα και επανειλημμένο σε μια αρνητική συμπεριφορά που, εναντί της οποίας είναι δύσκολο κανείς να αμυνθεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση της, της σεξουαλική παρενόχληση την ορίζει ως μη αρνητική συμπεριφορά σεξουαλικής φύσεως που μπορεί να είναι ε, σωματική, ε, λεκτική ή μη λεκτική ε, με στόχο ή αποτέλεσμα την αξιοπρέπεια της, του ατόμου. Και αυτές οι δράσεις έχουν μεγάλο πλάτος μπορεί να ξεκινάμε μέχρι το, από το το σεξισμό ε, και να φτάνουμε μέχρι τη μισογενία κλπ. Ε, η, η τάση όμως είναι να περιοριστούν οι ορισμοί. Θα ξανάρθουμε σε αυτό το θέμα αργότερα. Τώρα, τι θέλουμε να συστήσουμε. Χρειάζεται ένας ενιαίος ορισμός για την παρενόχληση και τον bullying σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή, παρόλο που οι ερευνητές συγκλίνουν, αυτή τη στιγμή έχουν πολλούς ορισμούς ακόμα. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη σεξουαλική παρενόχληση, θα πρέπει να ακούσουμε τις γυναίκες για να καταλάβουμε καλύτερα τι νιώθουν αυτές ότι είναι σεξουαλική παρενόχληση. Και να χρησιμοποιήσουμε τις δική τους φωνή ο, για να δώσουμε τον πιο κατάλληλο ορισμό και να καθαρίσουμε τα όρια του τι είναι και τι δεν είναι παραδεκτή συμπεριφορά. Και γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε και ένα πιο προσεκτικό λεξιλόγιο. Δεν μπορούμε όλες τις καταγγελίες να τις θεωρήσουμε σεξουαλική παρενόχληση. Εκεί θέλουμε να έχουμε διάφορους βαθμούς σοβαρότητας των πράξεων. Ε, μιλάμε για δείκτες ε, και εδώ έχουμε ορισμένες από τις χώρες που έχουμε στον πίνακά μας. Ε, τα αποτέλεσματα αυτά βασίζονται σε έρευνες ε, χίλιων ατόμων σε κάθε χώρα ε, σε, συγγνώμη, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης και βλέπετε τις διαφορές μεταξύ του 2015-2010 έχουμε μια σχετική αύξηση στις περισσότερες περιπτώσεις. Αυτό που θέλω να υπογραμμίσω είναι αυτό που είπε και η συγγήτρια. Κοιτάζοντα κοιτάζοντας τις ευρωπαϊκές χώρες θα δούμε περισσότερα, αρκετά ψηλότερα νούμερα στις βόρειες και δυτικές χώρες και πιο χαμηλά ποσοστά Στι χώρε τη Ανατολική Ευρώπης και στου χώρου του Νότου. Θα το σχολιάσουμε και αυτό. Καταρχήν, ε, παρενόχληση στο χώρο εργασία. 5-10% του εργατικού δυναμικού έχουν υποστεί ε, τέτοιου είδους παρενόχληση, τουλάχιστον μια φορά. Σεξουαλική παρενόχληση, τα νούμερα είναι πιο αβέβαια. Ορισμένες έρευνες δείχνουν πολύ χαμηλά νούμερα, 1, 2, 3%. Αυτό όμως που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερος με το κίνημα MeToo, αποκαλύπτονται πολύ ψηλότερα νούμερα από όσα εκτιμώνται παλαιότερα. Χρειάζεται λοιπόν να γίνει καλύτερη μελέτη. Θα επανέλθω σε αυτό. Σε ό,τι αφορά τα υψηλότερα ποσοστά σε χώρες της Βόρειας και Δυτικής Ευρώπης, είναι ένα ζήτημα που έχει σχέση πιο πολύ με τη συνειδητοποίηση. Το είπε και η συγγήτρια ότι είναι θέμα πιο πολύ συνειδητοποίησης και ανεκτικότητας. Δεν υπάρχει κανένας λόγος που να δικαιολογεί λιγότερη παρενόχληση χώρες του Νότιας Ευρώπης. Το αντίθετο ενδεχομένως. Επίσης, είναι ενδιαφέρον το ότι η σεξουαλική παρενόχληση δείχνει να είναι σημαντικό πρόβλημα σε χώρες με μεγάλους δείκτες ισότητας των δύο φύλων, όπως για παράδειγμα στη Σουηδία. Ε, η ισότητα λοιπόν δεν εξαλείφει αυτομάτως το πρόβλημα. Ποιοι επηρεάζονται. Η σεξουαλική παρενόχληση είναι κυρίως πρόβλημα των γυναικών και ιδιαίτερα των νέων γυναικών. Όμως, νέες μελέτες δείχνουν ότι όλο και περισσότεροι άντρες δηλώνουν να υφίστανται τέτοιου είδου συμπεριφορά επίσης. Ναι, ε, λεσβίες, ε, γκέι, ΛΟΑΔ γενικότερα και άτομα με αναπηρίες ε, αντιπροσωπεύονται σε μεγαλύτερο ποσοστό στα αποτελέσματα. Τώρα, ε, τι προηγείται της ε, παρενόχλησης στον χώρο εργασίας. επηρεάζεται το, η παρενόχληση από διάφορους παράγοντες, οργανωτικούς και, περι, και ε, εργασίας. Για παράδειγμα, σύγκρουση ρόλων, ε, η, ο τρόπος με τον οποίο ασκείται η, εξουσία των ηγετών, των επικεφαλής, το για παράδειγμα, πολύ συχνά όταν ο επικεφαλής ε, είναι πολύ χαλαρός, αυτό οδηγεί σε αύξηση του ποσοστού και, και εκεί που οι, οι ξέρουν να χειρίζονται το προσωπικό, ε, μπορούν να λειτουργήσουν ως buffer, ως προστασία έναντι της, ε, παρενόχλησης. Χρειάζεται λοιπόν ισχυρή, ισχυρά ηγετικά προσόντα. Το θέμα της κατάχρησης εξουσίας έχει άμεση σχέση με τη σεξουαλική παρενόχληση. Το έχουμε πει επανειλημμένως. Δεν πρόκειται για πόθο, σεξουαλικό πόθο, αλλά για κατάχρηση εξουσίας. Επιπλέον, ε, είναι πολύ σημαντικό να δούμε και την ανοχή της σεξουαλικής παρανόχλησης. Είναι ένα σημαντικός παράγοντας. Εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανεκτικότητα βλέπουμε και μεγαλύτερη κατάχρηση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις συνέπειες της παρενόχλησης, Είναι σαφές ότι το πρόβλημα είναι σοβαρό. Η ηθική παρενόχληση ε, αποτελεί κοινωνικό στρες που επηρεάζει την υγεία των ατόμων. Γι' αυτό υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες, έρευνες 25-30 ετών. Σε σχέση με άλλα φαινόμενα στον χώρο είναι από αυτά που δημιουργούν πραγματικό μετατραυματικό ε, ε, ε, δημιουργούν μετατραυματικές ασθένειες κλπ. Επίσης, επηρεάζει, μάλλον, η, η προσωπική αντοχή αποτελεί δίχτυ προστασίας. Αλλά αν αλλά αυτό μόνο για μικρής κλίμακας και έντασης ε, παρενόχληση. Όταν πολύ συχνά κανείς εκτίθεται σε τέτοιου είδους ε, συμπεριφορές, ε, μπορεί τα αποτελέσματα να είναι εξίσου αρνητικά. Μερικοί είναι πιο ευάλωτοι, άλλοι λιγότερο. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά τελικά, αν η πίεση, η έκθεση είναι επανειλημμένοι, ο καθένας θα υποστεί τις ίδιες συνέπειες. Και οι λιγότερο και οι περισσότερο ευάλωτοι. Επίσης, είναι, σημαντικά, είναι σημαντικό το οργανωτικό κόστος. Ε, έχουν το, η, η παρενόχληση επηρεάζει πάρα πολύ το, ε, την επίδοση, ε, την, α, την αδικαιολόγητη απουσία των εργαζομένων και γενικότερα το έργο που προσφέρουν οι υπάλληλοι στο χώρο εργασίας. Ε, επηρεάζεται δηλαδή η επίδοση όχι μόνο των ίδιων των υπαλλήλων που υφίστανται την παρενόχληση, αλλά και των υπολείπων στο ίδιο γραφείο, στην ίδια επιχείρηση. Συστάσεις. Χρειαζόμαστε περισσότερο επιστημονικές ε, μελέτες που να βασίζονται σε περισσότερα δεδομένα, πιο ασφαλή, θα έχουν πιο ασφαλή ε, για τη φύση και τη διάδοση του φαινομένου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης περισσότερες μελέτες ό,τι αφορά τις ανδρικές εμπειρίες σεξουαλικής παρενόχλησης. Για να δούμε αν διαφέρουν αυτές από τις εμπειρίες των γυναικών. Πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη ε, σημασία στην συνύπαρξη σεξουαλικής και ηθικής παρενόχλησης. Τώρα ιδιαίτερα που οι γυναίκες μπαίνουν σε καινούριου χώρους εργασίας, για παράδειγμα ε, στο στρατό και αλλού. Πολύ συχνά εκεί αυτά τα δύο φαινόμενα συνυπάρχουν. Και για τους άντρες βέβαια, αλλά ιδιαίτερως για τις γυναίκες. Επίσης, χρειαζόμαστε μελέτες που θα εξερευνούν την εμπειρία προστατευόμενων ομάδων. Έχει γίνει λόγος για το ζήτημα των διακρίσεων πως νεο, νεότερα άτομα, άτομα προέρχονται από εθνοτικές μειονότητες, άτομα ΛΟΑΔ ή άτομα με αναπηρίες, πώς αυτά αντιμετωπίζουν αυτό το φαινόμενο, σε ποιο εύρος κλπ. Πολύ συχνά είναι πολύ ψηλά ως σχετικά ποσοστά στα νούμερα μας. Σε ό,τι αφορά το δημόσιο χώρο, παραδοσιακά όταν μιλάμε για παρενόχληση και στο παρελθόν όταν μιλούσαμε για σεξουαλική των γυναικών, υπογραμμίζαμε το τι γίνεται σε απομονωμένα μέρη, μη δημόσιους χώρους δηλαδή. Τώρα οι έρευνες δείχνουν ότι στους δημόσιους χώρους παρουσία πολλών άλλων ατόμων, η σεξουαλική παρενόχληση επίσης συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό. Κάτι που σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουμε ε, εστίαση η παρενόχληση σε δημόσιους χώρους ε, είναι πολύ πιο διαδεδομένη. Ε, το 25% των γυναικών λέει ότι έχει υποστεί σεξουαλική παρενόχληση σε δημόσιο χώρο. Αυτό έχει σχέση με το γεγονός ότι τίνουμε να συνηθίσουμε στο φαινόμενο αυτό, να το θεωρούμε φυσιολογικό, να ε, μπανάλ. Επίσης θα πρέπει να συνδεθεί η σεξουαλική παρενόχληση σε δημόσιους χώρους με τη σεξουαλική παρενόχληση αλλού. Δηλαδή τα λιγότερο σοβαρά παραπτώματα σχέση με τις γυναίκες συνδέονται και με τα πιο σοβαρά. Δηλαδή υπάρχει ο σεξισμός, υπάρχει η μισογενία κλπ. που υποτίθεται ότι είναι λιγότερο προσβλητικέ πράξει, και πολύ συχνά όμω συνδέονται με πολύ πιο σοβαρά παραπτώματα και αδικήματα. Υπάρχει και ένας πολιτιστικός, μια πολιτιστική διάσταση Ε, σχόλια για το πώς ε, είναι μια γυναίκα, πώς έχει ντυθεί, πώς είναι ντυμένη κλπ. Ε, σε ορισμένες χώρες, σε ορισμένες κουλτούρες θεωρούνται πολύ πιο φυσιολογικά, πολύ πιο παραδοσιακά και πολύ πιο ανδρικά χαρακτηριστικά. Η, η σεξουαλική παρενόχληση επίσης πολύ συχνά συνδέεται και με την κατανάλωση αλκοόλ με την υπερβολική κατανάλωση τα όρια απαλήφονται και ο καθένας πιστεύει ότι μπορεί, έχει το δικαίωμα να κάνει περισσότερα πράγματα από ό,τι έχει. Συστάσει αυτό το θέμα, σε αυτό το τομέα. Χρειάζεται να συζητηθεί δημοσίως για το θέμα ε, της, ε, του ότι θεωρείται ε, κατά κάποιο τρόπο φυσικό φαινόμενο και αποδεκτό φαινόμενο. πολύ συχνά σεξουαλικά, σεξουαλική παρανόχληση γίνεται σε δημόσιους χώρους και πολύ συχνά γυναίκες λένε ότι ε, εντάξει τι να κάνουμε, συμβαίνει αυτό ε, ε, στα μπαρ όταν πίνουν οι νέοι κλπ. Και, ε, και πολύ συχνά επίσης δεν καταγγέλλονται τέτοιου περιστατικά. Επίσης την ιδέα ότι οι γυναίκες έχουν δικαίωμα να παρελοχλούν τις γυναίκες αναζητώντας σεξουαλική ικανοποίηση. Αυτό θα πρέπει να αμφισβητηθεί δεν είναι τμήμα της σεξουαλικής απελευθέρωσης αυτό το φαινόμενο, παρόλο που ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού θεωρεί πως είναι. Θα πρέπει να αμφισβητηθεί αυτή η τοποθέτηση. Χρειάζεται μια πιο σφαιρική προσέγγιση. Να δούμε πώς οι αξίες και οι κουλτούρες μιας κοινωνίας ε, ε, συχνά προωθούν την ανισότητα και τη βία εναντίον των γυναικών και πώς η βία σε ένα τομέα επηρεάζει την ε, βία σε άλλους τομείς. Και όταν λέω τομέα εννοώ σφαίρα, σφαίρα η, η οικιακή σφαίρα, η βία στην οικιακή σφαίρα επηρεάζει και το πώς ε, συμπεριφέρονται οι άνθρωποι δημοσίως, στη δημόσια σφαίρα, στο δημόσιο χώρο. Τώρα, στην πολιτική ζωή. Λίγο πίσω παρακαλώ. Σε ό,τι αφορά τον πολιτικό βίο και εκεί έχει συζητηθεί μέσω της εκστατείας του. Εδώ βλέπουμε τον μισογυνισμό και το sexual harassment πολύ διευρυμένα, πολύ διαδεδομένα, όπου συνδυάζονται και με πολιτιστικά ή με την πρόσληψη σε πολιτικές θέσεις και πίεση για να συγγύσουν. Αν θέλω δηλαδή να συνεχίσω την πολιτική μου σταδιοδρομία, τότε κατά κρατήσω το στόμα μου κλειστό. Αυτό λένε στο θύμα. Και συχνά σε τέτοιε περιπτώσει δεν θέλουν καμιά φορά οι γυναίκε ή τα θύματα να ευλάψουν το πολιτικό του κόμμα μέσα σε ε, μια πλανημένη αίσθηση πολιτικής ε, πίστης σε ένα κόμμα ή μια ιδεολογία. Οι συμπεριφορές λοιπόν δεν αμφισβητούνται και το γεγονός ιδιαίτερα ότι οι συμπεριφορές υψηλά ισταμένων πολιτικών, οι οποίοι καταφέρουν να ξεφεύγουν από τις ε, ενδεχόμενε συνέπειες του ε, γενετήσιου harassment. Και δημιουργείται έτσι και καλλιεργείται μια ε, κουλτούρα σιωπής. Το μη του εξέθεσε πολιτικούς σε πολλές χώρες που έχουν κάνει τέτοια πράγματα για χρόνια, ακόμα και σε βόρειες χώρες όπως οι σκανδιναβικές, όπου πολιτικοί ηγέτες και πολιτικά κόμματα ε, αναγκάστηκαν οι πολιτικοί ηγέτες ή και άλλοι, δηλαδή αναγκάστηκαν να απαρατηθούν από τα αξιώματά τους πράγματα, τα οποία γνωρίζαμε από χρόνια, αλλά κανένας δεν έκανε απολύτως τίποτα κατά αυτόν. Συμβαίνει επίσης ότι ορισμένοι πολιτικοί οι ίδιοι μπορούν να είναι θύματα bullying ή sexual harassment από μέλη του κοινού. Είδαμε και επιθέσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπου ορισμένοι θεώρησαν ότι ήταν πολιτικό bullying. Αυτές οι καταχρηστικές πρακτικές σε, μέρη, μέρος των μέσων μπορεί να είναι και μέρος της πολιτικής ζωής, έχουν όμως πάρα πολύ αρνητική ε, επίπτωση στη συμμετοχή γυναικών στο πολιτικό ε, γίγνεσθε. Ανοχή σε έντονες αλλά πολιτισμένες συζητήσεις και επιχειρήματα πρέπει να αναμένεται μεταξύ πολιτικών και βεβαίως και στο πώς αντιμετωπίζουν το προσωπικό τους. Ορισμένοι πολιτικοί όμως ε, παρανοούν, νομίζουν ότι η εκφοβιστική χρήση της γλώσσας είναι πολιτικός λόγος. Δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον ίδιο τρόπο γλώσσα στους ίδιους τους υφισταμένους σου ή στα μέλη του προσωπικού σου. Βλέπουμε και μάλιστα σε ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακόμη οι πολιτικοί έχουν πρόσβαση σε πολλαπλές πηγές και πρέπει να δεχθούν ότι υπάρχει ένα, είναι υψηλά ο πύχης για το τι ε, θα πρέπει να δέχονται ως κριτική του κοινού. Από την άλλη μεριά, βέβαια, εάν απομονώνονται κάποια άτομα για τις απόψεις τους με τρόπο που να προκαλείται μίσος, κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται να γίνεται ανεκτό. Πρέπει να εξευρεθεί μια ισορροπία ανάμεσα σε μια έντονη δημόσια πολιτική συζήτηση και στο τι μπορεί να είναι ανεκτό μέσα στα πλαίσια αυτά. Οι ψηλά επίπεδα ε, προσβολών και μίσους στα μίδια καμιά φορά θεωρείται ε, ε, αποτρέπουν ανθρώπου από το να διαλέξουν μια πολιτική σταδιοδρομία και ιδίω γυναίκες. Πώς αντιμετωπίζετε λοιπόν το bullying και η σεξουαλική παρενόχληση. Ας δούμε πρώτα τον τόπο εργασίας. Οι ευρωπαϊκές ρυθμίσεις δίνουν ξεκάθαρα μηνύματα και προβλέπουν και κάποια ε, βασική ε, κατεύθυνση. Αν δούμε τώρα τις ε, νομοθεσίες διάφορες χώρες μέλη, δεν υπάρχει ενιαία προσέγγιση για το bullying και για το sexual harassment. Ποικίλουν από χώρα σε χώρα και συχνά εντάσσονται μεταξύ των διατάξεων υγιεινής και λοιπά, καμιά φορά σε θέματα διακρίσεων και αλλού. Ενώ όμως οι ρυθμίσεις αυτές ασφαλώς δίνουν κάποια σημαντική νομοποίηση στην σοβαρότητα των θεμάτων αυτών, η αποτελεσματικότητά τους στις επιμέρους χώρες είναι αβέβαια και χρειάζονται περισσότερες μελέτες ακόμη για να εξεταστούν αυτά. Υπάρχει ένα ας πούμε νέο πλαίσιο, βεβαίω έχει ήδη μια ε, ηλικία 10 ετών, που λέγεται Framework Agreement για Harassment και Violence at Work από τους Ευρωπαϊκούς Κοινωνικούς Εταίρους. Αυτό εγκρίθηκε το 2007 και περιλαμβάνει και αυτή τη συμφωνία πλαίσιο, η οποία έγινε αντικείμενο διαπραγμάτευσης από τους κοινωνικούς εταίρους στην Ευρώπη, δηλαδή εργοδότες και εργαζομένους, οργανώσεις δηλαδή των ΜΕΝ και των ΔΕ και μετά από μακρές διαπραγματεύσει κατέληξε σε μια καλή συμφωνία η οποία εισήχθη και υπογράφηκε σε πολλέ χώρες μέλη. Ωστόσο, δυστυχώ είναι άγνωστο σε πολλού ανθρώπου ακόμη και αυτό είναι κρίμα. Πολλοί εργοδότες έχουν ε, εισαγάγει πολιτικές με τοπικά πρότυπα συμπεριφοράς για να δώσουν τη δυνατότητα καταγγελιών και επανόρθωσης. Δεν είναι πάντοτε αποτελεσματικά τα μέτρα αυτά, ιδίω διότι χωλαίνει η δέσμευση των ε, μάνατζερ. Όταν εξετάζουμε τις συστάσεις στον χώρο αυτό, όπως είπα, πρέπει να τονίσουμε και πάλι τη σημασία του, της συμφωνίας πλαισίου, που μπορεί να αποτελέσει έναν τρόπο ώστε μη συνδικαλισμένοι οργαζόμενοι να έχουν υποστήριξη. Υπάρχει και μια εναλλακτική επιλογή, υπάρχει οδηγία για την ηθική και σεξουαλική παρενόχληση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία μπορεί να προσφέρει στήριξη σε μεμονωμένους ε, απασχολουμένους. Σημαντική είναι επίσης η εμπιστευτικότητα σε περιπτώσεις ε, bullying και sexual harassment. Η ανωνυμία όμως Ιδίω σε σχέση με το Me όπου ορισμένοι καταγγέλθηκαν χωρίς την δυνατότητα να υπερασπιστούν αυτούς, θα πρέπει να αποφεύγεται η ανωνυμία. Όποιος ε, καταγγέλλεται ή ε, κατηγορείται για κάτι θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Οι καταγγελίες θα πρέπει να διαρευνώνται αντικειμενικά και χωρίς καθυστέρηση από τους ανθρώπους που θα έχουν τις αναγκαίες ε, ικανότητες. Και χρειαζόμαστε βέβαια και μια ε, γλώσσα με περισσότερες αποχρώσεις για τα σχετικά αδικήματα. Πολλοί άνθρωποι είπαν ότι ε, δεν θέλουν να καταγγέλουν περιστατικά σεξουαλική παρενόχληση δεν θεωρούν ότι είναι αρκετά σοβαρά τα επεισόδια αυτά, διότι ο τρόπο με τον οποίο ερμηνεύουν την σεξουαλική παρενόχληση ορισμένε οργανώσει, τα αρεβάζουν σε τόσο σοβαρό επίπεδο που το αποτέλεσμα είναι ότι θα χάσουν τη δουλειά του οι, οι η συγκεκριμένη συμπεριφορά. απλώ να υποστεί ο δράστης ένα πειθαρχικό Ενδεχομένω να υποστει ο δραστη ενα πειθαρχικο μετρο αλλα να έχει τη δουλειά του και ο ένα και ο άλλο σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση τώρα του bullying και του sexual harassment στο δημόσιο χώρο, ε, λίγη πρόοδος έχει γίνει με την προτινόμενη ε, Ευρωπαϊκή Οδηγία. Εμείς θεωρούμε ότι εκστατείες κατά της ε, βίας κατά των γυναικών, όπως η εκστρατεία MeToo, δεν επιτυγχάνουν τους στόχους τους. Νόμοι κατά του Τη παρενόχλησης ε, στο δημόσιο χώρο, στο δρόμο, έχουν εισαχθεί σε ορισμένε χώρες όπως Βέλγιο και Πορτογαλία με αβέβαιη αποτελεσματικότητα. Επίση είναι σημαντικό να διώκονται ποινικά σεξιστικέ ε, δράσει, ε, όπως τα σφυρίγματα. Αυτό προβλέπεται στη Γαλλία. Υπάρχει το πρόβλημα επίσης του χαμηλού επίπεδου επιτυχιών και της επιβάρυνσης του θύματος. Όταν λοιπόν μιλούμε για νέα μέτρα, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι έχουμε και τους αναγκαίους πόρους, για παράδειγμα αστυνομικέ δυνάμεις, για να ασκήσουν τις διώξεις. Όταν λοιπόν προτείνεται όπως στη Γαλλία ε, επιγραμμική καταγγελία, θα πρέπει να υπάρχουν, επαναλαμβάνω, οι αναγκαίοι πόροι. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι υπάρχουν Ξαναλέω, η αναγκαίοι πόροι. Χρειάζεται και μια ευαισθητοποίηση σε συνδυασμό με εντονότερη αστυνομική παρουσία για να δώσει θετικά αποτελέσματα. Είδαμε για παράδειγμα σε δημόσια φεστιβάλ στην Ισπανία όταν συζητήθηκε το θέμα αυτό ε, με το κοινό ε, με ταυτόχρονη όμως αστυνομική παρουσία η ανοχή του σεξισμού και της σεξουαλικής παρενόχλησης είναι ζήτημα πολιτιστικό το οποίο πρέπει να ξεπεραστεί. Είναι συχνά ταμπού ακόμη μεταξύ των νέων ανθρώπων και θα πρέπει να αρχίσει να συζητείται ήδη από τα σχολεία. Τώρα το bullying και το sexual harassment στην πολιτική ζωή. Υπάρχουν κατευθυντέ γραμμές για τους ευρωβουλευτές μεταξύ αυτών και μηχανισμοί για την αντιμετώπιση ε, ε, ακατάλληλης συμπεριφοράς από τα μέλη και από το προσωπικό με αμφισβητούμενη αποτελεσματικότητα. Λίγα εθνικά κοινοβούλια των χωρών μελών και πολιτικοί θεσμοί έχουν ε, αναπτύξει κατευθυντήρες γραμμές και πολιτικές για την συμπεριφορά. Αρχίζει και αλλάζει όμως αυτό. Ήδη ένας αριθμός χωρών αρχίζουν να, εισάγουν σχετικούς κώδικε. κώδικες. Και αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν και διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης πολιτικά κόμματα δεν μπορούν να αυτοαστυνομευθούν. Οι πολιτικοί θεσμοί δεν θα πρέπει να αναμένουν από τα πολιτικά κόμματα να αυτοαστυνομεύονται. Θα χρειαστεί διαμεσολάβηση, η οποία καμιά φορά επιτυγχάνει σε περιπτώσεις bullying και κυρίως στις πρώτες φάσεις αρνητικής συμπεριφοράς κατά κάποιων ανθρώπων. Με άλλα λόγια, είναι απολύτως λάθος ο δράστης ε, να προσπαθεί να έρθει σε διαπραγμάτευση με το θύμα για να, δουν αν υπάρχει, να δουν αν υπάρχει κάποια. Αντιθέτως θα πρέπει να ε, ε, επιβάλλονται κυρώσεις στον ε, δράστη. Μου μένουν δύο διαφάνειες. Έχω κάποια σχόλια για την συζήτηση περί μη του. Υπάρχει αυτή η αιμονή του προβλήματος σε χώρες λίγο πολύ παντού και όχι μόνο σε ορισμένες περιοχές. Άρχισαν να συζητούν θέματα όπως ε, στους κύκλους της τέχνης ε, των ε, μέσων κλπ. Αλλά όμως η εκστρατεία μη του έδειξε ότι το πρόβλημα υπάρχει παντού, στα σχολεία, στους δρόμους, σε, όλες, σε όλα τα επαγγέλματα. Υπάρχει διαφωνία για το εάν θα πρέπει να κατανομάζονται δημοσία άνθρωποι που κάνουν τα πράγματα αυτά ή αν θα πρέπει κυρίω ε, να στοχεύσουμε στο τι συμβαίνει σε βάρο των γυναικών. Υπάρχουν σημαντικέ διαφορέ ε, στάσεω μεταξύ διαφόρων χωρών και χωρών που έχουν πολλέ ομοιότητε μεταξύ του κατά τα άλλα. Για παράδειγμα, μεταξύ Σουηδία και Δανία, οι Σουηδοί φαίνονται να είναι πιο αυστηροί απέναντι στο sexual harassment, ενώ οι Δανείοι φαίνεται να είναι πολύ πιο ανεκτικοί. Και μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας, όπου η Γαλλία φαίνεται να είναι αυστηρότερη από την Γερμανία. Να έρθω στα συμπεράσματα. Υπάρχει ανάγκη για να γίνει αυτή η συζήτηση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίω για τα όρια του αποδεκτού και τη αξιοπρεπού συμπεριφορά. Τι ακριβώ σημαίνει sexual harassment και, και τι σημαίνει non-sexual harassment. Πρέπει λοιπόν να συζητηθεί και να ζητηθεί τι ενδεχομένω είναι ανεκτό και τι όχι χρειάζεται να οριοθετηθούν τα λιγότερο σοβαρά αδικήματα και τα πιο σοβαρά. Και το γεγονός ότι η συμπεριφορά σε ένα χώρο επηρεάζει τη συμπεριφορά και σε άλλους. Πρέπει να αντιμετωπιστεί το bullying και το harassment ως πολιτιστικά, πολιτιστικές εκδηλώσεις και εκεί να αναλυφθεί η δράση σε πολλαπλά επίπεδα με μια συνολική απάντηση που να λαμβάνει υπόψη και την πρόληψη και την παρέμβαση ότι αν συμβαίνει κάτι, όταν κάποιος δηλαδή υφίσταται bullying ή sexual harassment και την επανόρθωση και του θύματος αλλά και της οργανώσεως. Και χρειάζεται, υπάρχει χώρος για συλλογική δράση. Θα πρέπει να είναι καλοδεχούμενη η συλλογική δράση, διότι η ανεκτικότητα και η αντιμετώπιση ως ομαλής μιας τέτοιας συμπεριφοράς είναι από τους μεγαλύτερους εχθρούς και γι' αυτό χρειάζεται να ζητήσουμε από τις γυναίκες να διατηρήσουν την πίεση επί των πολιτικών θεσμών και της κοινωνίας στο σύνολό της ώστε να αλλάξουν οι πρακτικές αυτές. Thank uh, Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε καθηγητά για την παρουσίασή σας. Βεβαίως που είναι πολύ χρήσιμο αυτά που ακούσαμε. Και τώρα να ακούσουμε την κυρία Πιτσένο, την ε, εισηγήτρια. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ιδιαίτερως να ευχαριστήσουμε τον καθηγητή για την ε, σφαιρική, πλήρη, ε, παρουσιασή του και όλα αυτά θα είναι πάρα πολύ χρήσιμα για το έργο το οποίο έχουμε να επιτελέσουμε τις αμέσως επόμενες μέρες. Σας ευχαριστούμε. Ελπίζω να συνεχιστεί η συνεργασία μας. Σας ευχαριστούμε για όσα κάναμε και ευχαριστώ όμως και τους συναδέλφους για όσα είπαν που είναι σημαντικά. Οπότε ελπίζουμε τελικά το έργο μας να είναι εις όφελος των ε, γυναικών και έτσι να σταματήσουμε το φαινόμενο αυτό της βίας. Κυρία Ζαμπόσκα. Πολύ σύντομα, Πρόεδρε. Ο καθηγητής μας είπε ότι η μελέτη αυτή κακώς προσιάζεται από κάποιον ηλικιωμένο και ότι θα έπρεπε να παρουσιάζεται ε, από κάποια νέα γυναίκα. Όχι. Ε, τα, τα θύματα είναι γυναίκες. Ναι, θα έπρεπε να έχουμε κάποια γυναίκα. Αλλά θα έπρεπε και οι άντρες να είναι πρωτοπόροι στην σε αυτού του αρνητικού φαινομένου. Γι' αυτό και τελικά είμαι ευχαριστημένη μας το προσφύγει ο καθηγητής γιατί χρειάζεται νομοθεσία, χρειάζονται συμφωνίες πλαίσιο. για την κοινωνία είναι απαράδεκτο και το bullying και η παρενόχληση. Μηδενική ανοχή. Αυτή είναι η σωστή προσέγγιση για το αρνητικό φαινόμενο. Πολλές φορές η κοινωνία παίρνει το μέρος του ενόχου, του υπέτειου παρενόχλησης και όχι του θύματος. Μην το ξεχνούμε αυτό. Θα πρέπει να υπάρχει σεβασμό τη ε, αξιοπρέπεια, οπότε τότε πια να είναι πυρητική η νομοθεσία. Ευχαριστούμε κυρία Ζαμπόσκα, ευχαριστούμε κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ όλου. Λήξη τη συνεδρία Όχι. Συνεχίζει η πρόεδρο. Και τώρα. Mm. Α, ήθελε το λόγο. Α, συγγνώμη, συγγνώμη κύριε καθηγητά. Φοράει τα φυσικά και ο καθηγητή. Εδώ δώσω το λόγο στην συναδελφόλη θέλω να σας πω ότι δεν θα έχουμε διερμηνία μετά τις μία. Μέχρι τις μία διερμηνία. Μετά θα αποχωρήσουν οι διερμηνίες. Ευχαριστούμε την ομάδα των ερευνητών για την εξαιρετική δουλειά που έκαναν μέσα από την έρευνα που μας παρουσιάσαν σήμερα. Αργήσαμε να συζητήσουμε ανοιχτά για την εξασφαλική παρανόχληση και το εκφοβισμό στο χώρο εργασίας. Έπρεπε φαίνεται να ξεσπάσει σκάνδαλο για να αποφασίσουμε να μιλήσουμε ανοιχτά και στο δικό μα σπίτι. Με σοκάρει το γεγονό πω το πιο δημοκρατικό υποτίθεται όργανο τη Ευρωπαϊκή Ένωσης έχουμε υψηλά ποσοστά παρενόχληση. και θέλω να τονίσω πως δεν μιλάμε μόνο για σεξουαλική παρενόχληση και ούτε πρέπει να μας ενδιαφέρει μόνο αυτή τη μορφή επειδή είμαστε η Επιτροπή Γυναικών. Δεν υποθυμώ φυσικά καθόλου αυτή τη μορφή, αλλά οι γυναίκες ως ευάλωτη ομάδα είναι και πιο συχνά θύματα της ψυχολογικής και ληκτικής παρενόχλησης που δυστυχώς δημιουργούμε και εμείς οι βουλευτές οι υψηλά αισθαμενοι επειδή έχουμε περισσότερη δύναμη. Διαλύει τους η παρενόχληση, τη ζωή και την αξιοπρέπειά τους. Σχετικά με τα μέτρα που προτείνει η μελέτη, πρόληψη, αλλαγή νοοτροπίας και πολιτικής, δημιουργία κανόνων και κυρώσεων, ας πάρουμε τον οδικό χάρτη που υιοθετείται του Προεδρείου του Ευρωκοινοβούλιο και ας βάλουμε ημερομηνίε στα μέτρα που πρέπει να υιοθετηθούν. Αγαπητές, αγαπητοί συνάδελφοι, ο ρόλος μας δεν θα πρέπει να είναι απλώς να κάνουμε άλλη μια κοβέντα, αλλά να παρακολουθούμε συνεχώς αν τα, αν τα πραγματοποιηθούν τα μέτρα που υιοθέτησε το Προεδρείο του Ευρωκοινοβουλίου. Έχουμε ήδη κατηστηρίσει πάρα πολύ. Δεν αρκεί να λέμε πώς θα στηρίξουμε τη Συμβουλευτική Επιτροπή, να τις φέρουμε άμεσως εξωτερικός ε, εξειδικευμένος και πυρογνώμονες να βάλουμε από τώρα χρονοδιάγραμμα για υιοθέτηση κώδικα ευπρεπούς συμπεριφοράς και κυρώσεων. Μας έχει μείνει ένας χρόνος ως το τέλος της θητείας. Αν δεν έχουμε υιοθετήσει κανόνες έως τότε, στη νέα θητεία θα πρέπει να αρχίσουμε πάλι από την αρχή και στο μεταξύ να υπάρχουν άνθρωποι που τα συνεχίζουν να υποβάλλονται σε αυτή την απαράδεκτη μείωση της αξιοπρέπειας και της προσωπικής τους προσωπικότητά τους. Και τα είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι αυτό. Ευχαριστώ. Thank you, Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Κούνεβα. Ευχαριστώ. Αυτό ήταν το τελευταίο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Σας ε, ενημερώνω ότι η επόμενη συνάντηση θα είναι στις 14 και 15 Μαΐου. Ευχαριστώ όλες και όλους την γραμματεία, η ευχαριστή και τους διερμηνείς και εσάς κύριε καθηγητά.